τους ομιλητές πέρα της ε, συζήτησης. Αύριο στις 12 η σχετική ψηφοφορία. Και τώρα, στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, την έκθεση ΕΣΑΙΑ για τις τεχνικές απαιτήσεις για τις μεταφορές πίστοσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ. Καταρχάς, η κυρία Βόρτμαν Κόλ έχει το λόγο. Όντω uh, uh, Όντως, κύριε Πρόεδρε, δεν περιμένατε να μιλήσω εγώ, αλλά δυστυχώς ε, τα προβλήματα στο αεροδρόμιο του Σχίπχολ, ε, ειδοποίηση για βόμβα, ε, απέτρεψαν την κυρία Εσάγια από το να έρθει στην ώρα της. Μου ζήτησε λοιπόν να μιλήσω εκ μέρους της. Εξ ονόματος της λοιπόν θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα του τρομερούς διαλόγου και από τη συμφωνία με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους ε, του Συμβουλίου, τον Επιτρόπο Μπαρνιέτε, τον κυρία Μπόλς από την Επιτροπή Νομισματικών Υποθέσεων, τους κοιόδες εισηγητές και όλους όσοι υπέβαλαν τροπολογίες και συνέβαλαν σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα και ασφαλώς και στην γραμματεία της Επιτροπής Οίκων. Η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Χώρου Πληρωμών σε ευρώ είναι πάρα πολύ σημαντική και έχει πάρα πολλά πλανεκτήματα για τους πολίτες. Από τον Φεβρουάριο του 2014 όλες οι ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι εξίσου εύκολες όσο και πληρωμές σε μετρητά. Πολλούς θα ωφελήσει αυτό, αλλά προφανώς θα είναι ε, δυνατόν να γίνουν πληρωμές από όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς προς όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη. Και οι μεταφορές πιστώσεων θα αντιμετωπίζονται σαν εγχώριες μεταφορές. Θα χρησιμοποιείται μόνο ένας ε, ε, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, μίας μορφής, το IBAN, και αυτό θα έχει πολλά πλανεκτήματα, θα χρειάζεται για όλο τον ευρωπαϊκό χώρο με ένας μόνο λογαριασμό. Ακόμα και αν το άτομο δουλεύει σε άλλο κρατό μέλος. Μπορεί, για παράδειγμα, να έχει τη μισθοδοσία του σε λογαριασμό στη χώρα του. Και έτσι θα μπορεί να χρησιμοποιείται και μία ενιαία πιστοτική κάρτα σε όλον τον ενιαίο χώρο πληρωμών. Όταν, για παράδειγμα, πάει κανείς διακοπές, θα μπορεί να επωφελείται από όλα αυτά τα ωφέλη. Αυτό αποτελεί καλή είδηση για το ευρώ και για την ε, ευρωζώνη. Θα ανοίξει τον ανταγωνισμό, θα καταστήσει τις πληρωμές πιο βοηθητικές. Και θα αποφέρει 123 δισεκατομμύρια σε περίοδο εξαετίας. Και τα ωφέλη αυτά θα είναι ακόμα πιο σημαντικά, γιατί αυτός ο χώρος πληρωμών θα ευνοήσει τις καινοτομίες, όπως για παράδειγμα η παράλληλη σύνδεση, όπως γίνεται στη Φιλανδία και στην Ολλανδία, με το λογιστικό σύστημα των ε, υπηρεσιών, των επιχειρήσεων, οι εύκολες πληρωμές επίσης ε, καταστούν και πιο εύκολες τις αγορές μέσω διαδικτύου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι καταναλωτές θα μπορούν πραγματικά να συγκρίνουν τις τιμές και να βρίσκουν την καλύτερη τιμή. Η αγορά ενός υπολογιστή από τον πιο φτηνό πάροχο μπορεί να ρίξει τις τιμές παντού στην εσωτερική αγορά. Άρα, από πολλές απόψεις, ε, αυτός ο ευρωπαϊκός χώρος πληρωμών είναι πάρα πολύ σημαντικός για μια εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική αγορά. Ως τώρα ήταν πολύ βραδύ ρυθμοί, ρυθμή ανάπτυξης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις ε, κατάφερε να πετύχουν να πετύχει την ίδια προθεσμία και για τις άμεσες ε, χρεώσεις και για τις μεταφορές πιστώσεων. Φεβρουάριο του 2014 και για τα κράτη-μέλη που δεν έχουν, δεν χρησιμοποιούν το ευρώ, ε, η ημερομηνία αυτή θα είναι ε, Οκτώβριος του 2016. Αυτό θα είναι εύκολο, θα διευκολύνει μάλλον τις ε, εκστρατείες πληροφόρησης των πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης πέτυχε το σωστό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει από την τράπεζα να περιορίσει την συλλογή πιστώσεων και επίσης δεν θα χρειάζεται ο καταναλωτής να δίνει στην τράπεζα την ιδιαίτερο κώδικα, κωδικό BIC μετά από δύο χρόνια. Ούτε καν για διασυνοριακές πληρωμές για την καλύτερη προσαρμογή στο νέο σύστημα. Υπάρχουν κάποιες εξαιρείες σε διετούς ε, μεταβατικής περίοδου. Για παράδειγμα, κάποια κράτη-μέλη, ένα κρατός μέλος, για παράδειγμα, μπορεί να επιτρέψει στις ε, τράπεζες για δύο χρόνια να μην χρησιμοποιεί την, το σταθερό μορφότυπο XML ή να χρησιμοποιεί για μεταβατική φάση δύο ετών το παλιό μορφότυπο του λογαριασμού. Κύριε Πρόεδρε, η οδηγία θα, η σχετική οδηγία θα αναφερθεί αργότερα μέσα στο έτος και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να οριστικοποιηθεί το σύστημα στο σύνολό του και προκειμένου να καταστεί εύρυθμο. Εξ ονόματος της κυρίας Σάγια θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι χαιρόμαστε και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλη σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο πληρωμών που πλέον ε, οι άμεσες χρεώσεις και μεταφορές πιστώσεις μπορεί να γίνουν σαν κανονικές εγχώριες ε, πληρωμές. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο Μπαρνιέ. Merci, Madame la ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή ε, Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, την Πρόεδρό της κυρία Μπόλους και η κυρία Βόρτμαρ Κόλλα. Σας παρακαλέσω να διαβεβάσετε στην κυρία Σάρια Σαγιά τις ευχαριστίες μου για την εργασία που έκανε σε πολύ Καλή συνεργασία με τους ε, σχεδόν ηγητές, την κυρία Ιντβέλτε, Γκίγκολτ και η Βαρή Μπαντάρ. Οι υπηρεσίε πληρωμών είναι ε, πολύ σημαντικέ για τι οικονομίε μα, γιατί αν δεν λειτουργούν σωστά, δεν μπορούμε να έχουμε εσωτερική αγορά που να παράγει όλο αυτό το δυναμικό συναλλαγών ε, υπέρ της ανάπτυξης. Ο κανονισμός που είναι υποσυζήτηση θέλει να υλοποιήσει το ΣΕΠΑ. Ε, δηλαδή τον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ. Το πρόγραμμα ΣΕΠΑ θέλει να αναπτύξει τις υπηρεσίες πληρωμών σε ευρώ, να μην είναι πια κατακαιρματισμένες από μια χώρα σε άλλη, αλλά κοινέ για το σύνολο της Ένωσης και να αντικαθιστούν τις ε, υπηρεσίες χώριων ε, πληρωμών. Είναι μάλιστα το παράδειγμα μιας τέτοιας οικονομικής ρύθμισης στην υπηρεσία των νόσων που βρίσκονται μέσα στην πραγματική οικονομία να γίνουν οι διασυνορικές πληρωμές τόσο εύκολες όσο και οι εγχώριες με μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία για τους πολίτες στην υπηρεσία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ε, θα υπάρχει μεγαλύτερο ανταγωνισμό σε αυτό το τομέα και άρα πιστεύω πως θα μειωθεί το κόστος των πληρωμών, πράγμα που θα, μάλλον θα πρέπει επίσης να ενισχύσει την καινοτομία. Και να χαιρετήσω εδώ και μια πρόοδο σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Είναι μια νέα απόδειξη της πραγματικής χρησιμότητας της εργασίας που κάνουμε. Το είπατε και εσείς κυρία Βόρτμαν Κόλ, ειδικά τη στιγμή της, του τριμερού διαλόγου και με, μεγάλη μου χαρά Διαπιστώνω πως τα κείμενα της Κομισιόν βελτιώνονται και διευκρινίζονται χάρη στις εργασίες του Κοινοβουλίου. Σε έκθεση της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής της κυρίας Εσαγιάς συνέβαλε τα μάλα στη βελτίωση της πρότασής μας. Ε, είναι ακόμη, περισσότερο, ακόμη πιο ευνοϊκό για τους καταναλωτές πρώτον γιατί λόγω της προγραμματισμένης ε, ε, εξάλληψης του κώδικα BIC από το 2016 δηλαδή μια λιγότερη πληροφορία για να κάνει κανείς με πληρωμή είτε πρόκειται για χώρα είτε για διεθνή. Δεύτερον, η κατάργηση του επιπλέον κόστους για κάθε διασυνοριακή πληρωμή και αυτό από τη στιγμή που θα αρχίσει να ισχύει ο κανονισμός. Βεβαίως, εμείς ε, ε, δεν ε, είμαστε ευχαριστημένοι λόγω της ε, κατάρρησης των διαφορετικών ημερομηνιών για την μεταφορά των πληρωμών ή των πιστώσεων γιατί για μας θα διευκόλυνε περισσότερο τις επιχειρήσεις. Ωστόσο και μια ενιαία ημερομηνία θα μπορούσε να διευκολύνει τη μετακίνηση προς το ΣΕΠΑ και τη χρήση των νέων αριθμών λογαριασμού IBAN. Ε, είμαστε λοιπόν ικανοποιημένοι για την τελική συμβαστική λύση. Είμαστε έτοιμοι να ασχοληθούμε με τη διακυβέρνηση του ΣΕΠΑ μέχρι το τέλος του 2012, όπου θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος, και καθώς και επίσης για το θέμα των δικαιωμάτων του καταναλωτή μέσα στο πλαίσιο της αναθεωρημένης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών. Αυτές οι δύο, σε αυτά τα δύο σημεία έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο δηλώσεων αρχής με βάση τις ε, εξ, ε, αρμοδιότητες της Κομισιόν και αυτά βρίσκονται στο παράρτημα που σας έχει υποβληθεί και αντικατοπτρίζουν λέξη προς λέξη τη συμβιβαστική στην οποία φτάσαμε το Δεκέμβριο. Τέλος, ε, κυρία Πρόεδρε, με αυτόν τον κανονισμό δίνουμε στην αγορά πληρωμών ένα νομικό πλαίσιο το οποίο χρειάζεται. Συμβάλλουμε στην ανάδυση ενός πραγματικού μιας πραγματικής αγορά, ενιαίας αγοράς πληρωμών και Έχουμε μια νέα αγορά πλέον όπου οι πληρωμές θα γίνονται σε ολόκληρη την Ένωση τόσο γρήγορα, τόσο αποτελεσματικά όσο και στο ε, εσωτερικό ε, χάρη σε αυξημένο ανταγωνισμό με χαμηλότερο κόστος. Αυτό είναι το τρίτο σημείο που συζητάμε από το απόγευμα. Πρόκειται για μια συγκεκριμένη πρόοδο για την εσωτερική αγορά υπέρ των πολιτών και των επιχειρήσεών μας. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Εύελιν Γκέπχαρτ εξ ονόματος Επιτροπής Καταναλωτή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Καταναλωτή ασχολήθηκε με το θέμα του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ, του ΣΕΠΑ, γιατί εδώ τίθεται ένα θέμα προστασία του καταναλωτή και πρέπει να πω ότι είμαι ικανοποιημένη με το συμβασμό που εξαιρέθηκε, γιατί κάποια από τα θέματα τα οποία έχει αποφασίσει η Επιτροπή μα αποτυπώνονται στην έκθεση. Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό για το ότι μπορούμε να πούμε στους καταναλωτές ότι και εδώ στην ενιαία αγορά σκεφτόμαστε τον καταναλωτή. Αυτή η εντύπωση δεν είναι πάντα ιδιαίτερα έντονη. Τα όρια σε ό,τι αφορά τις μεταφορές πληρωμών αποτελούν όρια στην Ευρώπη. Σύνορα. Είναι στα σύνορα. Θα πρέπει λοιπόν να ξεπεραθούν, να ξεπεραστούν και να μην εμποδίζουν την κινητικότητα. Και χαίρομαι που σε ό,τι αφορά την μεταφορά των πληρωμών. Στο μέλλον όλες οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές ε, θα μπορούν με ένα λογαριασμό σε μια οποιοδήποτε χώρα να διεξαγάγουν τις εργασίες τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ιδιαίτερα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι μόνο για αυτές, αλλά και για καταναλωτές οι οποίοι μετακινούνται ιδιαίτερα ή βρίσκονται σε διακοπές. Είναι πολύ θετικό το ότι φροντίσαμε να υπάρχει ένα ενιαίο, ενιαίο χρονικό σημείο μεταφοράς ε, και σε ό,τι αφορά και τις ε, μεταφορές. Ε, δεν θα ήταν καλό για τους καταναλωτές να υπάρχουν δύο χρονικά σημεία, δύο προθεσμίες. Αυτό θα προκαλούσε ίσα ίσα πιο πολύ σύγχυση. Νομίζω ότι η σαφήνια και η νομική βεβαιότητα είναι τα ζητούμενα. Και αυτό είναι που πετυχαίνουμε και με την έκθεση αυτή. Ένα τρίτο και τελευταίο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι το εξή. Η πληροφόρηση των πολιτών και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί φοβούνται αυτό το IBAN γιατί θεωρούν ότι έχει πάρα πολλούς αριθμούς. Αν καταλάβουν όμως, αν κάποιος τους πει από τι αποτελείται, δεν είναι καθόλου δύσκολο, δεν είναι καθόλου περίπλοκο. Μία ενημερωτική εκστρατεία για να ξέρει ο πολίτης τι αντιμετωπίζει. Θα περάσουμε τώρα στους ομιλητές εξ ονόματος των ε, πολιτικών ομάδων. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Γκέι Μίτσελ πρέπει να λάβει το λόγο, αλλά επειδή δεν είναι στην αίθουσα, θα ζητήσω από τον συνάδελφο Ιβάρη Παντάρ, από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, να πάρει το λόγο. Συνάδελφοι, πρώτα πρώτα επιτρέψατε μου να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, διότι με επιτέλεσε έργο πάρα πολύ αξιόλογο. Επίσης, να ευχαριστήσω και όλους τους κοιόδης εισηγητάς, διότι πρόκειται για μια έκθεση που είναι παράδειγμα προς μίμηση. Φαίνεται πως η κοινοτική μέθοδος έτσι μας πηγαίνει σε κάποια αποτελέσματα πάρα πολύ θετικά, προοδευτικά, τα οποία προωθούν το ιδεώδες της ενιαίας κοινή αγορά διότι ε, ήταν κάτι που χρειαζόταν αυτή η ρύθμιση για τις πληρωμές. Το, το δε χάος το οποίο ε, κυριαρχούσε από καιρού καιρών, διότι ο καθένας και του δικού του κανόνες αυτό ήταν κάτι το οποίο παρέβλεπτε το, το, το εμπόριο, παρέβλεπτε την κοινή αγορά. Παρέβλεπτε. Και οπότε θα έπρεπε να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση την εναρμόνιση των διαφορετικών συστημάτων να βρεθεί μια συμβαστική λύση. Βεβαίω, όλε οι αλλαγέ έχουν το τίμημά του και χρειάζεται πάντοτε χρόνο ρονταρίσματο. Και πάντω για του σοσιαλιστέ και δημοκράτε η αφετηρία ήταν αυτή η αναγκαιότητα για κάποιου κοινού ευρωπαϊκού κανόνε. Επίση όμω, τονίζουμε το ότι ε, θα χρειαζόταν να προστατεύσουμε τους ε, καταναλωτάς αλλά και κάποιες ε, αποτελεσματικές πρακτικές. Θα πρέπει φυσικά να φραγωστεί διόντως ο νόμος αλλά να, να σας ε, να σας τονίσω το ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά ε, τις τιμές, το τι γίνεται σε περίπτωση που ο ανταγωνισμός εντείνεται, οπότε θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαγγελνίζει τέτοιε περιπτώσει για το οποίο θα ισχύσει και αμέσω μόλι θα θέσει ισχύ ο εν λόγω κανονισμό. Η δε διαχείριση αυτών των συστημάτων ήταν κάποτε προνομίο των τραπεζών. Τώρα, θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι όμω να συμμετάσχουν στη διαχείριση και την εποπτεία. Ακόμη, η κώδικε. εντομισμού, δεν θα χρειαζόταν πλέον για τι ιστορικές πληρωμές από τον Απρίλιο του 2014, αλλά και για τις ιστορικές πληρωμές από το Φεβρουάριο του 2016. Επίση. από ε, το, το, το, το πρότυπο των, των εμβασμάτων από το τοπικό, από το τοπικό φορμάτ στο διεθνές, στο ΙΜΠΑΝ είναι κάτι το οποίο θα εφαρμοστεί, γιατί είναι, είναι λογικό επίσης θα υπάρχει μία μεταβατική περίοδος για τις πληρωμές. Ε, οπότε μπορείτε να δείτε τώρα τι, πώς, πόσο ωφελεί το να καταβάλουν προσπάθειες από κοινού και πώς όλοι ωφελούνται. Οπότε, ακριβώς λόγω αυτού του ΣΕΠΑ, ε, θα ωφεληθεί όλος ο κόσμος. Μιλάμε για μια εξαιτία 120 τόσα δις ευρώ. Είναι επομένω ένα παράδειγμα προβλήματο και ελπίζουμε να δούμε περισσότερε δράσει τέτοιε στο μέλλον. Να δώσω το λόγο στην κυρία Σοφία Ιντβέλτ από την ομάδα των Φιλελευθέρων. Yes, thank you, Chair. Κυρία Νετφέλτ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και πρώτα πρώτα να ευχαριστήσουμε το, την εισηγήτρια η οποία παρά τα προβλήματα που πρέπει στο αεροδρόμιο δεν μπορούμε παρά να γνωρίσουμε αυτό το οποίο ε, επετέλεσε. Να δούμε επομένω τι έγινε όσον αφορά όλα αυτά τα, τα, τα θετικά που θα προκύψουν, όπως είπε ο εκπροσωπών την εισηγήτρια, αυτά τα ΣΕΠΑ έχει ε, στα ελληνικά, θα πρέπει να δούμε σε ποιο διαδικασία θα οδηγήσουν, να κάτσουμε να δούμε τι πλεονεκτήματα θα προκύψουν. Ε, όμως είναι κατανόητο. Γιατί? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ε, πήρε τόσο πολύ, γιατί θα πάρει τόσο πολύ, γιατί θέλει τόσο τόσες εξαιρέσεις, γιατί πήρε τόσο χρόνο να το εφαρμόσουμε και άλλο τόσο να το εφαρμόσουμε οριστικά ε, αφού τώρα σοβεί αυτή η κρίση. Βλέπουμε ότι μια τέτοια σχετικά μικρή προσπάθεια όσον αφορά αυτέ τι μεταφορέ πιστώσεων και αυτές, αυτά τα εμβάσματα ε, βλέπουμε πόση ώρα χρειάζεται για να επιτελεστούν τότε καταλαβαίνουμε. Τότε καταλαβαίνουμε γιατί ο κόσμο θα πρέπει να μάθει και να συνηθίσει τα νέα συστήματα. Όμω, τι ζητάμε από του ε, Έλληνε συμπολίτε μα, Για κοιτάξτε τι έγινε στην Αραβική Άνοιξη. Τότε, για καθίστε και σκεφτείτε τα όλα αυτά. Αν, αλλάξουν, αν αλλάξει απλώ το φορμάτ του, του, του λογαριασμού, πάει το έμβασμα, τι θα γίνει αυτό, θα φέρει την αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, συμπαθάτε με, η, η, η Ευρώπη θα πρέπει να αλλάξει. Να αλλάξει στη ίδια αγορά για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τη θέση που θέλουμε στον κόσμο. Διότι ε, οι πληρωμέ είναι το, το, το, το, το καύσιμο για να τρέξει η κοινή αγορά. Και άρα θα πρέπει οι καταληκτικέ ημερομηνίε που είναι πάρα πολύ γενναιόδορε να τυπηθούν από τα κράτη-μέλη. Μιλάμε εδώ και για, για νέε μεθόδου. Βλέπουμε ότι θα υπάρξει μια διαδικασία που θα είναι ταχυτέρα μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ κυρία Ιντβέλτ. Ήθελα τώρα να παρακαλέσω τον κύριο Σβέν Γκίγκολτ από την ομάδα των Πρασίνων να πάρει το λόγο. Ja, Frau Präsidentin. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ καταρχάς ε, για την καλή συνεργασία και μαζί σας κύριε Παρνιέ, γιατί φυσικά απότερο στόχος της έκθεσης είναι η Ευρώπη να καταστεί και μια ευρωπαϊκή, ε, ένας ευρωπαϊκός χώρος πληρωμών, ένας ενιαίος χώρος πληρωμών. Θα πρέπει όλα αυτά να διαμορφωθούν από κοινού, γιατί όπως είπε η συνάδελφος Σοφίν Φέλτ, όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν πραγματοποιηθεί πιο γρήγορα και στην περίπτωση αυτή αυτό θα είχε ωφελήσει και τους καταναλωτές πιο γρήγορα, αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θα έπρεπε να έχουν καθυστερήσει τόσο πολύ σε ό,τι αφορά την τήρηση των σχετικών προδιαγραφών. Τι θα γίνει τώρα με το σχετικό δίκαιο ανάκτησης, επιστροφής. Εμείς ως Κοινοβούλιο θέλουμε όλα αυτά να περάσουν απαραίτητος. Αυτό που είναι σημαντικό όμως είναι τα σχετικά δικαιώματα επιστροφής να παραμείνουν σε εθνικό επίπεδο, γιατί αυτό αποτελεί τη βάση για ένα χάος, αν θέλετε, που δεν θα προκληθεί, που αποφεύγεται στη Γερμανία και είναι σημαντικό ότι το Κοινοβούλιο πέτυχε το ηλεκτρονικό σύστημα στη Γερμανία να μπορέσει να περάσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τέλος, είναι σημαντικό και στο θέμα της ε, μεταφοράς πιστώσεων, να δεθούν το θέμα της δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ που συμφωνήσατε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών να μην αποτελεί την μοναδική πηγή προδιαγραφών, αλλά και αυτό να υπάγεται στον τομέα της δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ανυπομονώ και προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία. Λόγω στον κύριο Νίκο Χουντή από την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, η συζήτηση που κάνουμε ενδεχομένως μοιάζει να είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ενδεχομένως αυτή η εκτίμηση να προκύπτει από τον επηρεασμό που έχω από τις χτεσινέ αποφάσεις που με δραματικές συνθήκε έλαβε το ελληνικό κοινοβούλιο. μια λιτότητα ύφεση που βεβαίω δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. συζητάμε λοιπόν τη μεταβίβαση τη πληρωμής σε ευρώ σε μια περίοδο που η κρίση σοβεί η ύφεση βαθαίνει η λιτότητα αγκαλιάζει πολύ μεγαλύτερα κομμάτια της ευρώπης και μοιάζει ηρωνικό να λέμε ότι πρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα τη στιγμή που ενδεχομένω οι ευρωπαίοι πολίτε και οι ευρωπαίοι λαοί να μην έχουν ευρώ στην τσέπη του. απέτηση αυτού του συστήματος του ενιαίου χώρου και άμεσα ωφελημένοι προφανώς είναι οι αγορές τα χρηματοπιστωτικά συστήματα οι πολυεθνικές εταιρείες δική τους απέτηση ήταν να προχωρήσει αυτό το σύστημα. παρά τα αυτά επειδή πρέπει να προστατεύσουμε μέσα σε αυτό το κλίμα τα δικαιώματα των καταναλωτών οι παρατηρήσεις μου είναι πρώτον επειδή αυτό το σύστημα η αλλαγή που θα γίνει θα είναι πολυδάπανη και το κόστος θα είναι μεγάλο θα πρέπει το κόστος αυτό να μην το πληρώσουν οι πολίτες κατά τη γνωστή λογική που μεταβιβάζουν τράπεζες τέτοια κόστη προς τους πολίτες. η έκθεση δεν το καλύπτει. δεύτερον θα πρέπει να γίνει συστηματική προσπάθεια ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών. τρίτον και ιδιαίτερα σημαντικό επειδή θα αφορά και σε ηλεκτρονικό χρήμα θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα που δεν τα εξασφαλίζει η έκθεση από περιπτώσεις απάτης σε βάρος των καταναλωτών. θεωρώ θετικό ότι υπάρχει μια ημερομηνία θεωρώ θετικό ότι καταργήθηκε η διατραπεζική ε, χρέωση και πρέπει αυτό να γίνει και για τις κάρτες. σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Χουντή, ε, υπάρχουν δύο συνάδελφοι που έχουν ζητήσει να σας υποβάλουν ε, ερωτήσεις με τη διαδικασία της ε, μπλε κάρτας. Πρώτα θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Χάνς Πίτερ Μάρτιν. Παρακαλώ, κύριε Μάρτιν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μου προκάλεσε έκπληξη αυτό που είπατε στην αδελφή Χούντι πριν από λίγο. Η Ελλάδα είναι τόσο απομονωμένη που δεν έχει εμβάσματα στο εξωτερικό. Δεν αντιμετωπίζετε το πρόβλημα στο μέλλον ότι στο μέλλον θα υπάρχουν πάρα πολλοί υπηκοοί σα που θα βγουν στο εξωτερικό και θα δουλεύουν ε, σαν γκάσταρμπάιτρ και θα κάνουν βάσματα. Και όταν λέτε ότι δεν θα μπορέσουν να υποφεληθούν οι τράπεζες, δεν βλέπετε ε, ότι με την ενοποίηση αυτή θα υπάρχει ένα επιπλέον κέρδος ε, στις τράπεζες που θα μειωθεί, δηλαδή σε ό,τι αφορά τα εμβάσματα. Κύριε Χουντή. Απαντώ στο τελευταίο ερώτημα, μάλλον δεν έγινε σωστή κατανόηση της, ε, αυτό που είπα. Θα ωφεληθούν οι τράπεζες, δεν το αρνούμε. Επομένως, μάλλον για παρεξήγηση πρόκειται. Για τα άλλα που είπατε κύριε Μάρτιν, δεν τα αρνούμε. Αλλά θέτω το θέμα στην πραγματική βάση ή τουλάχιστον αν θέλετε τις παρατηρήσεις σε ποια περίοδο ζούμε και αν υπάρχουν εισοδήματα ή μάλλον περικόπτονται αυτά τα εισοδήματα και επομένως υπάρχει η ουσία σε ποια οικονομική κατάσταση ζούμε σε ποια οικονομική κατάσταση βρίσκεται η ευρωπαϊκή ένωση. αυτό δεν μπορείτε να το αρνηθείτε φαντάζομαι και δεν αφορά μόνο την ελλάδα ότι αυτή η ύφεση και η λιτότητα περιορίζει τα εισοδήματα. από εκεί και πέρα όπως είδατε στο θέμα αυτό υπησήλθα σε παρατηρήσεις που τούτων δοθέντων μπορούν να το βελτιώσουν. Κύριε Γκίγκολτ, θέλετε να θέσετε ένα ερώτημα. Uh, Αγαπητέ συνάδελφε, εγώ θέλω να σου θέσω μια ερώτηση μόνο. Αισθάνομαι πλήρη αλληλεγγύη με τους φτωχούς στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή πληρώνουν το κόστος της κρίσης. Ε, αισθάνομαι την ευθύνη και αισθάνομαι και συνυπεύθυνος για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ολόκληρος. Αυτό που δεν καταλαβαίνω όμως είναι ότι έκανες, κάνατε πολύ συγκεκριμένα ε, παρατηρήσεις για τις αλλαγές στο ΣΕΠΑ. Δεν σε είδα όμως στις συναντήσεις δεν σας είδα, δεν είδα τους, ε, το επιτελείο σας και ήθελα να ρωτήσω εδώ γιατί θέτετε ερωτήσεις ενώ μπορούσατε και είχατε τη δυνατότητα να υπερασπιστείτε τις θέσεις σας εκεί στην Επιτροπή. Χρησιμοποιείτε διπλή γλώσσα. Νομίζω ότι ο κύριος συνάδελφος δεν χρησιμοποίησε σωστή ορολογία για πολλού και διαφόρου λόγου ενδεχομένω δεν μετήχα στι διαδικασίε για να πω την πρώτη γνώμη. Άρα δεν με συλλάβατε σήμερα να λέω δεύτερη γνώμη. Και δεύτερο, κύριε συνάδελφε, οι παρατηρήσει είναι πάρα πολύ συγκεκριμένε και νομίζω ότι η Ολομέλεια μα επιτρέπει να κάνω παρατηρήσει επί τη εκθέσεω που δεν με περιορίζει κανένα, δεν ξέρω γιατί εσεί πρέπει να με ελέγξετε. Επομένω δεν υπάρχει διπλή γλώσσα, υπάρχουν οι παρατηρήσει οι οποίε είναι πάρα πολύ συγκεκριμένε. Ευχαριστώ κύριε Χουντή και τώρα θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Σαμ Ποτέρχο ε, εξ ονόματος της Ευρώπης Ελευθερίας και Δημοκρατίας. Σα arvoisa puhemies. Yhteinen euromaksualue. ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτός ο νέος χώρος πληρωμών σε ευρώ είναι μια καλή πρωτοβουλία. Πιστεύω πως είναι μια πρωτοβουλία η οποία στηρίχθηκε από τους πολίτες και κυρίως από τις επιχειρήσεις. Είναι πολύ πιο πρακτικό και μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα ίδια στοιχεία για τις πληρωμές παντού στην Ευρώπη και αυτό αφορά και την ηλεκτρονική χρέωση τα ηλεκτρονικά τιμολόγια είναι μια πολύ σημαντική βάση. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια πρακτικά προβλήματα. Για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι πιο αποτελεσματικές από ό,τι άλλες. Υπάρχουν αποφάσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή σε κάποιες χώρες. Ε, αν υπάρχουν άλλες που δεν έχουν, χώρες όμως που δεν έχουν θέσει εφαρμογή αυτέ τι αποφάσει και δεν έχουν, ε, δεν, δεν, τότε δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτέ τι εξοικονομήσει. Αυτό το σύστημα ε, δημιουργεί λοιπόν κάποια προβλήματα, μάλλον δημιουργεί προβλήματα για τις χώρες που το έχουν ιδιοθετήσει. Για παράδειγμα στη Φιλανδία είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε πολύ μακρές σειρές ε, αριθμών για τους λογαριασμούς και οι πολίτες ε, δυσκολεύτηκαν πολύ να αρχίσουν να χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα. Γιατί οι εσωτερικές μας πληρωμέ είναι τώρα το ίδιο δύσκολο με τις πληρωμέ ε, στο εξωτερικό. Πρέπει ωστόσο να βιαστούμε γιατί πρέπει να ενεργήσουμε. Για μένα η μετάβαση θα πρέπει να γίνει σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και όσο γίνεται πιο σύντομα. Τέλος ο κύριος Χάνς Πίτερ Μάρτιν από τους μη εγγεγραμμένους. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Μια παλιά απέτηση ε, αυτών που βρίσκουν τα διάφορα πράγματα έτσι πολύ κεντρικά και γραφειοκρατικά είναι πως στην Ευρώπη πρέπει κανείς να τη βλέπει στην καθημερινή τη ζωή. Ε, θεωρώ πως αυτό το οποίο κάνουμε είναι ένα κομμάτι ευρωπαϊκής άνοιξης. Η θερμοκρασία ανεβαίνει. Συναντά ένα τον άλλον. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ πέρα. και ως άμεσους βεβαίως εμείς ε, γείτονες έχουμε την ε, Γερμανία και την Ελβετία ξέρετε και ξέρετε μια φορά για να κάνω μια, ένα έμβασμα πέντε Υπάρχει ένα πρόβλημα με την ε, γαλλική μετάφραση Υπήρξε πρόβλημα με τη γαλλική διερμηνία, γι' αυτό χρειάστηκε να σας διακόψω. Συγγνώμη. Μπορείτε να ξεκινήσετε και πάλι την ομιλία σας. Ευχαριστώ. Δεν, μου είχε συμβεί, αλλά ευχαριστώ, δεν μου είχε συμβεί μέχρι τώρα. Αλλά ευχαρίστω να ξαναξεκινήσω. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι οι οποίοι ασκούν κριτική για εδώ πέρα συγκεντρωτισμό κτλ. Πρέπει να δουν πώς πράγματι ερχόμαστε ένας πιο κοντά στον άλλον και έχουμε πράγματι μια ευρωπαϊκή άνοιξη. Και έχω συγκεκριμένες εμπειρίες από τις δύο γειτονικέ μας χώρες και ιδίω σε, αυτές, σε αυτή την ε, χιλιετία γιατί μου είχαν γράψει ένα πρόστιμο στη Γερμανία από, πώς το λένε, από 5 μάρκα κατέληξε λόγω της καθυστέρησης να αυξηθεί στα 10 και με τα έξοδα του εμβάσματος κατέληξα να πληρώσω 70 μάρκα για ένα αρχικό πρόστιμο 5 μάρκων. Τώρα μπορούμε να το νιώθουμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Δεν κοστίζει τίποτα. Δεύτερον, πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις συναλλάσσονται με το εξωτερικό δεν το πιστεύετε, αλλά αυστριακές και με την Γερμανία και με την Τσεχία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και ε, βεβαίως ήταν σοβαρό το κόστος ε, του εμβάσματος. Μιλάμε για 0,25% το οποίο κατέβηκε ε, μετά από πολλές διαπραγματεύσεις και σε άλλε περιπτώσει ήταν και πολλά σοβαρότερα τα ποσά. Τι έκαναν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, κρατούσαν πολλού λογαριασμού σε διάφορε χώρε και βεβαίω ήταν πάρα πολύ δύσκολα μετά τα λογιστικά και τα βιβλία του Και αναποτελεσματική αυτή η κατάσταση. Είναι καλό λοιπόν αυτό το οποίο γίνεται τώρα, αλλά βεβαίω, πράγματι έπρεπε να έχει γίνει και πιο νωρίτερα αλλά είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση που νομίζω πως θέλουμε όλοι, δηλαδή να μπορούμε να βλέπουμε πιο ξεκάθαρα τι πώς έχουν οι ε, ροές, οι πληρωμές και γι' αυτό το επαναλαμβάνω χαίρομαι για να όταν έχουμε τέτοιες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στους άλλους εγγεγραμμένους ε, ομιλητές και πρώτα θέλω να παρακαλέσω τον Ζαν Πολ Γκοζές να πάρει το λόγο για δύο λεπτά παρακαλώ. Merci, Madame le Président. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Συνάπη, κύριε Επίτροπε. Ξέρετε πόσο εκτιμώ τις δράσεις σας, όλα όσα κάνετε. Το θέμα με το οποίο θα απόψε είναι σημαντικό. Ήμουν εισηγητή, ξέρετε, τη οδηγία για τι υπηρεσίε πληρωμών στην προηγούμενη θητεία και γνωρίζω πόσο η δουλειά για αναρμόνιση των υπηρεσιών των πληρωμών στην Ευρώπη είναι κάτι σημαντικό. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε κάτι το οποίο είναι ενοχλητικό η Πολυμερής ε, Επιτροπή Συναλλαγών. Από την αρχή επρασπίζομαι αυτή την ε, επιτροπή και είχα την ευκαιρία να το πω όταν ξεκινήσαμε την πρώτη μεταφορά σε ΠΑ το έτος 2007. επιτροπή, ε, οι επιτροπές αυτές είναι θεμητές. Αυτό που δεν είναι θεμητό είναι ο καθορισμός των ποσών όταν είναι υπερβολικά. Γιατί αυτές οι επιτροπές είναι διότι η υπηρεσία πληρωμών είναι κάτι εμπορικό και θα πρέπει τα ιδρύματα τράπεζα ή τρα, ίδρυμα πληρωμών που δημιουργείται από το κεφάλαιο 2 τη οδηγία που προανέφερα ε, έχουν, ασκούν εμπορική δραστηριότητα, άρα είναι κανονικό να έχουν μια αμοιβή. Αυτή η αμοιβή θα πρέπει προφανώς να δικαιολογείται από την παραχωρηθή υπηρεσία. Και από αυτή την άποψη η Επιτροπή σε αυτών των ε, συναλλαγών καθοριζόταν ε, ε, καταχρηστικά. Άλλαξαν τα πράγματα τώρα και η κατάσταση στην οποία βρίσκομαι με το νέο κείμενο, με το νέο κανονισμό είναι αρκετά παράδοξη. Πρώτα απ' όλα μέσω του κειμένου ρυθμίζουμε ένα θέμα το οποίο συζητείται και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εγκρίνονται οι επιτροπές συναλλαγών αυτός μέχρι το 2007 ε, για εθνικό επίπεδο και μετά σε διεθνές. Αλλά Όσον αφορά επίση απόρριψη πληρωμών, του επιτρέπουμε να λειτουργούν. Δεν είναι συνεκτικό. Δεν θα πρέπει αυτό που έγινε αυτή τη φορά να μπορεί να είναι ένα παράδειγμα για εκείνο που θα γίνει ε, για τι απόλυτε τραπεζικέ στι μελλοντικέ ρυθμίσει. Νομίζω ότι ο προβληματισμό θα πρέπει να διεξαχθεί καλύτερα στον τομέα και θα πρέπει βλέποντα ότι μόνο έξι επιτροπέ έχουν, μόνο έξι χώρε αυτέ τι επιτροπέ να πούμε την άχρηστο. Γιατί, Γιατί πρώτα απ' όλα διαφάνεια δεν υπάρχει, πληρώνουμε τι υπηρεσίε πληρωμών μέσω άλλου είδου αμοιβών, μέσω άλλων πόρων. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ. Θέλω να καλέσω στο βήμα τον συνάδελφο Κούτα για δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε Μπαρνιά, αγαπητοί συνάδελφοι, στηρίζω την πρόταση για τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς ε, πληρωμών σε ευρώ, διότι αυτό θα διευκολύνει σημαντικά το σύστημα το οποίο είναι στη διάθεση των Ευρωπαίων καταναλωτών. Οι καταναλωτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν μία ενιαία μέθοδο πληρωμής, ένα μόνο λογαριασμό για τις πληρωμές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την πρωτοβουλία αυτή θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των διασυνοριακών πληρωμών και η κατακαιρματισμένη αγορά θα γίνει ενοποιημένη. Ξέρετε ότι θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι από αυτό θα προκύψουν κέρδη πολλών εκατομμυρίων ευρώ ε, μέσα στην ε, επόμενη πενταετία εξαιτία λόγω των εξοικονομήσεων. Το θέμα είναι να δούμε τι ε, προθεσμίες υπάρχουν για τη μετάβαση προς ένα γενικευμένο σύστημα η μεταβατική διαδικασία, η μεταβατική περίοδος μάλλον δεν πρέπει να παραταθεί αδικαιολόγητα. Η αρχική στρατηγική η οποία είχε εγκριθεί σε σχέση με τις ε, μεταφορές πιστώσεων έλεγε ότι η μετανάστευση, η μετάβαση αυτά πρέπει να γίνει με βέλικτο τρόπο. Δεν κατέληξε όμως αυτό στα προεξοφληθέντα αποτελέσματα. Μόνο το 15,7% του συνόλου των εμβασμάτων στην Ευρωζώνη ε, γίνονται μέσω αυτού του Ευρωπαϊκού Συστήματος ε, Πληρωμών. Και νομίζω ότι είναι απαραίτητο επίση να εξασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών στη διάρκεια τη μεταβατική αυτή περίοδου. Εξού, κύριε Επίτροπε, σα συνιστώ να προβείτε σε κάποιε εκστρατείε ενημέρωση, πληροφόρηση, υποχρεώντα και τον τραπεζικό τομέα να συμβάλλει. Ε, ήθελα τώρα να παρακαλέσω τον κύριο Στογιάννο να πάρει το λόγο για 1,5 λεπτό, παρακαλώ. Λοιπόν, Μιλάμε για το θέμα της οικονομίας, όπου πληρωμές καταβάλλονται παραδοσιακά σε ευρώ, για ένα τομέα της οικονομίας, ο οποίος είναι η αγορά κινήτων, περιουσιών και ο τομέας των μισθώσεων. Όταν κάποιος θέλει να κάνει μία μεταφορά από βουλγαρική τράπεζα σε άλλη βουλγαρική τράπεζα αυτό θεωρείται σαν διεθνής μεταφορά αν αφορά ξένο νόμισμα και εισπράτεται ένα τέλος και στις δύο πλευρές της συναλλαγής. Αυτό είναι κάτι που αυξάνει κατά 10% το κόστος. Νομίζω ότι το έγγραφο το οποίο συζητούμε θα βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση, κυρίως για τις χώρες μέλη που είναι εκτός της Ευρωζώνης. Όμως υπάρχει και ένα άλλο θέμα, που είναι ανεξάρτητα από αυτά που συζητούμε για τα τέλη κλπ. που μπορούν να καθορίζονται από την αγορά. Η πρόταση που εμπεριέχεται στον κανονισμό δείχνει ότι Έχουμε νομικά μέσα για να ρυθμίζουμε τα τέλη και τις φορές. Αυτό το δρόμο θα πρέπει να ακολουθήσουμε στην Ευρώπη. Να πάρει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, μια κοινή εσωτερική αγορά απαιτεί ένα κοινό νόμισμα και ένα κοινό νόμισμα απαιτεί ένα χώρο πληρωμών. Η εφαρμογή αυτών των τριών στόχων βεβαίως γίνεται σε φάσεις και με δυσκολίες. Γι' αυτό σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω βρίσκεται σε συμφωνία με το Συμβούλιο. Πρώτη, ε, τέλος Φεβρουαρίου 2014 έχουμε την οριστική προθεσμία για την ολοκλήρωση της ζώνης ε, πληρωμών στην Ευρωζώνη και το 2015 για τις υπόλοιπες χώρες μη Ευρωζώνης. Δεν ε, είναι υποχρεωτικό να πάνε τόσο αργά τα πράγματα, αλλά βλέπουμε σήμερα πως ε, κάθε επιχειρηματίας πρέπει να ανοίγει λογαριασμό σε κάθε κράτος που δραστηριοποιείται. Ένας άνθρωπος ο οποίος ε, εργάζεται σε μία άλλη χώρα δεν μπορεί να πληρώνεται στην χώρα προέλευσής του. Θα μπορούσε να εξοικονομείται ένα ε, δισεκατομμύριο ευρώ. Γι' αυτό με τη σημερινή μας απόφαση ε, κάναμε πάρα πολύ μεγάλο έργο για τον καταναλωτή και για την προστέμενη αξία του να ανήκει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η κυρία Πρόεδρος και εγώ είμαστε συνυπεύθυνοι για το θέμα της επικοινωνίας. Και εδώ πέρα πρόκειται ακριβώς για ένα πολύ καλό παράδειγμα για το περί τίνος πρόκειται, τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κερδίζουν οι πολίτες. Δεν κάνουμε μόνο οικονομίες, διευκολύνουμε και την ζωή τους. Και βεβαίως διατηρείται έτσι η ε, παλαιά μορφή των παγίων εντολών, οι οποίες δεν θα πρέπει να αλλάξουν από εδώ και μπρος στο μέλλον. Ένας καλός συμβιβασμός. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μόνικα Φλασίκοβα Μπένιοβα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι, μια ενιαία αγορά με πληρωμές σε ευρώ χωρίς μεγάλες διαφορές μεταξύ των εθνικών συστημάτων είναι κάτι το απολύτως απαραίτητο για την λειτουργία της. Αυτά τα μέτρα πρέπει να έχουν ληφθεί εδώ και πολύ καιρό. Αλλά, αν βάση περιπτώσει, κάλιο αργά παραποτέ. Στο πλαίσιο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικαθίστανται τα διάφορα εθνικά συστήματα και έχουμε το ΣΕΠΑ, το Ευρωπαϊκό Σύστημα, το οποίο προσφέρει σε Ευρωπαίους καταναλωτές και επιχειρήσεις αξιόπιστες πληρωμές με ανταγωνιστικές τιμές. Πρόκειται λοιπόν για ευνοϊκές συνθήκες αύξησης του ανταγωνισμού και δυνατότητα γρηγορη εφαρμογής επιπλέον πρέπει νομίζω να έχουμε στο τέλος και οικονομίες και ε, αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος ε, και νομίζω πως θα οδηγηθούμε σε μειώσεις των ε, τιμών. Αυτό βοηθάει ιδιαίτερα εκείνες τις χώρες όπου αυτή τη στιγμή τα εμβάσματα είναι πάρα πολύ ακριβά. Αυτό έχει και πολιτικές πτυχές και είναι σημαντικό και για τη στρατηγική 2020 όπου θα γίνει πιο έξυπνη η λειτουργία της ε, οικονομίας και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μια γρήγορη μετάβαση στην ΣΕΠΑ. Ο ενιαίος αυτός χώρος είναι ένα καλό παράδειγμα της κοινοτική μεθόδου και όφελος των πολιτών. Τελευταίος εγγεγραμμένος ομιλητής, ο κύριος Ανδρέας Μέλτσερ. Η τεχνική πρόοδο και ο ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο πληρωμών έχει οπωσδήποτε μεγαλύτερα πλεονεκτήματα όσον αφορά την ρευστότητα και τους μικρότερους χρόνους των εμβασμάτων. Βεβαίω ε, θα πρέπει και και το ξέρουμε αυτό και οι κάρτες ε, να χρησιμοποιούνται όχι μόνο στα ATM αλλά και στα μηχανήματα αυτόματης χρέωσης των ε, λογαριασμών. Ε, τα πράγματα αυτά μπορούν να γίνουν αλλά δεν είναι τόσο απλά για να τα κάνουν όλοι και ειδικά οι ηλικιωμένοι. Γι' αυτό είναι καλό το ότι θα διατηρηθούν και οι παλαιοί αριθμοί λογαριασμών. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αυξάνεται η ηλεκτρονική εγκληματικότητα είτε μέσω επιθέσεων hacker είτε μέσω των υποτιθέμενων δωρεάν λογαριασμών όπου γίνεται ψάρεμα για να υποκλέψουν τα τραπεζικά δεδομένα, οπότε θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα υπαναχώρησης από τις ε, συναλλαγές αυτές, εάν μπορεί να αποδειχθεί πως δεν τις ήθελε ο χρήστης. Επίσης, θα είναι δυνατόν να γίνει η χρήση όλων αυτών των υπηρεσιών και από smartphone. Επίσης, θα πρέπει και οι τράπεζε να είναι σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν πιθανά προβλήματα με επιστοτικές κάρτες. Και πρώτα θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Σιλβέστρης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Αυτό που κάνουμε είναι άλλο ένα μεγάλο σημαντικό βήμα πρόοδου για ο τομέα των ιεών πληρωμών τη Ευρωζώνη με αυτή την ημερομηνία την 1η Φεβρουαρίου του 2014 είναι η ολοκλήρωση μιας αδρομής για την ενιαία αγορά και είναι ένα σημαντικό βήμα που ξεκίνησε σημαντικό βήμα για το ενίο νόμισμα. Είναι σημαντικό βήμα οικονομικό Υποθυμίζω στον Επίτροπο ότι, ε, ότι έγιναν οικονομίες, θα δικήσει οικονομίες ενός εκατομμυρίου σε σχέση με το σημερινό κόστος και είναι πολύ επωφελές για τον κατανοητή. Αυτή η ενία, ενίος χώρος πληρωμών σε ευρώ είναι ένα βήμα προόδου και το υπενθυμίζω αυτό στον Επίτροπο και το βλέπουμε θετικά. Είναι μια διαδρομή μέσω της κοινοτική ε, διαδικασίας ε, που είναι κάτι που ασθενίζεται το Κοινοβούλιο και η χώρα μου. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Σιλβέστρης και τώρα θέλω να παρακαλέσω την κυρία Τικάου να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Spațiul unic de uh, Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ είναι πολύ σημαντικός για την καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς Πρόκειται για ένα βήμα το οποίο προσφέρει την πλατφόρμα για την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Αν αυτό εγκριθεί σε ευρία κλίμακα θα ωφελήσει την μετάβαση των πληρωμών προς αυτό το σύστημα. Για να έχουμε όμως ωφέλη θα πρέπει τα πρότυπα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης να αντιστοιχούν ε, στα αντίστοιχα πρότυπα ISO. για τα μηνύματα που αφορούν τις ε, υπηρεσίες, τα οποία χρησιμοποιούνται. Θα πρέπει λοιπόν αυτά να ενταχθούν στο ε, σύστημα πληρωμών που ισχύει ε, για τα δημόσια, τους δημόσιους θεσμούς. Θα σας παρακαλούσα να μας δώσετε κύριε Επίτροπε κάποιες περισσότερες προφορίες. Μπασέσκου παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για εύρυθμη λειτουργία τη ενιά αγοράς η Ευρώπη χρειάζεται ένα σύστημα πληρωμών που να είναι ασφαλέ και αποτελεσματικό. Τα εθνικά προγράμματα δεν μπορούν να οδηγήσουν σε επαρκή όθηση για μια ταχεία μετάβαση και ολοκληρωμένη μετάβαση προς ενίο χώρο πληρωμών σε ευρώ. Το ΣΕΠΑ είναι το βασικό στοιχείο για τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς της υπηρεσίας των υπηρεσιών πληρωμών. Το ΣΕΠΑ θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους και θα επιτρέψει οικονομίες πάρα πολύ σημαντικές. Παραδείγματο χάρη, τα ενδεχόμενα κέρδη ωφέλη από το ΣΕΠΑ θα μπορούσαν να φτάσουν 400 δις ευρώ σε μία περίοδο εξαετή. Είναι σημαντικό να καθοριστεί μία τελική ημερομηνία κοινή για την αναρμόνιση των εισφορών και για τα εμβάσματα σε ευρώ είναι απαραίτητο ταυτόχρονα να ρυθμιστούν οι πολυμερείς επιτροπές συναλλαγών για το πώς θα καθορίζουν τις, τις εισφορές αυτές. Θα πρέπει να προωθηθεί το προϊόν σε πάλι, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ε, χωρίς να πέσουν τα σύνορα και στον τομέα των πληρωμών θα ήταν πάρα πολύ προβληματική. Γι' αυτό οι προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου πληρωμών με την δημιουργία διεθνών προδιαγραφών είναι κάτι το κατανοητό και κάτι το οποίο θα απλοποιήσει τις πληρωμές. Ε, το γεγονός πως ε, από το 2014 και οι χώρες Ευρωζώνης και από το 2016 οι υπόλοιπες χώρες ε, της ε, Ένωσης θα μπορέσουν να έχουν ενιαίες διαδικασίες ε, πληρωμών είναι ένα σημάδι για το ότι αυξάνεται και μεγαλώνει από κοινού η κοινή αγορά και οπωσδήποτε αυτό ωφελεί τους πολίτες μας και θεωρώ πως οι αλλαγές που θα επέλθουν στον τραπεζικό τομέα δεν θα αποτελέσουν εμπόδιο Eh, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική της δουλειά και για την ευεργετική αυτή απλούστευση του συστήματος πληρωμών χάρη σε αυτόν τον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ, ΣΕΠΑ. 23 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις σίγουρα θα χαρούν ιδιαίτερα ε, με τις καλύτερες αυτές ε, συνθήκες που δημιουργούνται και για ανάπτυξη και για εξοικονόμηση πόρων. Βέβαια χρειαζόμαστε μια πλατφόρμα ενημέρωσης για όλους. Και κάτι το οποίο σίγουρα χρειαζόμαστε επίσης είναι η αξιοπιστία διότι εν καιρό αποτυχίας τραπεζικών συστημάτων, εν καιρό διαδηλώσεων για, για τη Συμφωνία Άκτα, βλέπουμε ότι ενδέχεται να υπάρξουν ε, ταραχές και πρέπει να τους προσέξουμε. Στη διαδικασία Catch ο κύριος Τζέμκε. Αχα, ε, e, Από ό,τι κατάλαβα είναι η σειρά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Επίτροπε, έχω ερώτηση να σας κάνω. Πιστεύω ότι είναι αρκετά εύκολο ζήτημα αυτό για χώρες που ήδη έχουν το ευρώ σαν νόμισμα. Όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε και χώρες που θα ήθελαν να έχουν το ευρώ σαν νόμισμά τους. Έχουμε και χώρες οι οποίες είναι αρκετά συνεπείς και λένε ότι θέλουν να κρατήσουν το εθνικό τους νόμισμα. Εξού και ερώτησή μου, κύριε Επίτροπε. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι οι κανονισμοί που θα καλύπτουν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2016 και από ό,τι κατάλαβα θα τεθούν σε ισχύ την 31η Οκτωβρίου ενεστώτος έτος θα καλύπτουν και το Ηνωμένο Βασίλειο διότι γνωρίζουμε ότι το Ενωμένο Βασίλειο έχει τραπεζικό σύστημα που είναι σημαντικό για την Ευρώπη. Κύριε Μπαρνιέ, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω συγκεκριμένα στις ερωτήσεις ε, με όσο το πιο απλό τρόπο. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γκέπχαρτ η οποία επενθύμησε την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με το αρχικό κείμενο της Κομισιόν χάρη στο Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα δε σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών. Να πω στην κυρία Γκέπχαρτ αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους ότι σε ό,τι αφορά τις αιματοπιστωτικές υπηρεσίες Μία από τις μεγάλες προτεραιότητές μου για το έτος που ξεκίνησε το 2012 είναι η προστασία των καταναλωτών και θα το δείτε και στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας που ξέρει πολύ καλά ο κύριος Γκοζές για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, PSVM και τη διαμεσολάβηση μεσάζονται στις ασφάλειες. Και για το shadow banking θα κάνουμε μια πρόταση, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Βέβαια, αλλά τέλος πάντων η προστασία των καταναλωτών είναι προτεραιότητα. Και επειδή μιλάω για την προστασία των καταναλωτών και την πληροφόρηση, την ενημέρωση, να πω στον κύριο Κούτας και στον κύριο Παντά, στον κύριο Χουντή, στον κύριο Τερού. Είπε ένα από εσά ότι πρόκειται για ένα, μια αλλαγή. Πράγματι, για να τη διευκολύνουμε και να την επιταχύνουμε αυτή την αλλαγή, που είναι και πολιτισμική αλλαγή, πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και νομίζω ότι έχω δίκιο όταν λέω ότι και οι τράπεζε έχουν δεσμευτεί σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την εκστρατεία ενημέρωση. Και σε ό,τι αφορά τη μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία των καταναλωτών. Από στον κύριο ε, και στην κυρία Κόκοβιτ που πριν από λίγο μίλησε, ότι πραγματικά θα παρακολουθήσουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή την εφαρμογή του κανονισμού αυτού. Με τη μέρη που έχουμε να συνεργαστούμε με τις τράπεζες για την ε, σωστή υλοποίηση του προγράμματος. Φυσικά πρέπει να υπάρχει πολύ καλή διακυβέρνηση του συστήματος ε, του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ. Γιατί χρειάζεται τόσο χρόνος, ρωτήσατε, κυρία Ιντφέλτ. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε τα πράγματα να πάνε λίγο πιο γρήγορα. Συνεργασία Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και κομισιών, αυτή η συνεργασία των τριών θεσμικών οργάνων ε, είχε ίσως ε, ως αποτέλεσμα αυτή τη μικρή καθυστέρηση, αλλά θα ξεκινήσουμε. Υπάρχει αυτή η προσέγγιση το 2014 για την Ευρωζώνη, το είπε και ο κύριος Κάρας. Να πω και στην κυρία Τικάου επίσης ότι εδώ μιλάμε για ένα πραγματικό εργοτάξιο ε, που ξεκινά και επιταχύνεται για τον ε, νέο χώρο πληρωμών. Υπάρχει όμως και ένα ακόμη σχέδιο που ξεκινά και αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Να σας πω λοιπόν ότι εδώ έχουμε να επεξεργαστούμε θέματα άκρο τεχνικά, τα οποία αφορούν τον, την ηλεκτρονική τιμολόγηση, την ηλεκτρονική υπογραφή, την ασφάλεια των πληρωμών. Οι συνάδελφοι Νταλή και Κρός από την Κομισιόν ε, εξετάζουν με πολύ μεγάλη προσοχή όλους αυτούς τους ε, εμπορικούς ε, φραγμούς για να λύσουν τα προβλήματα. Ο κύριος Χουντής έκανε μια αναφορά την οποία κατανοώ λόγω της πάρα πολύ σοβαρής κατάστασης την οποία βιώνουν οι Έλληνες πατριώτες του. Σε αυτό το στάδιο όμως δεν θα ήθελα να επισέλθω ε, στη συζήτηση αυτή, ε, δηλαδή στις προσπάθειες που όλοι μας πρέπει να κάνουμε ε, για να υπάρξει ανάκαμψη και ανόρθωση της κατάστασης. Στην ε, χώρα σας, κύριε Χουτίτη, γνωρίζω και τη σέβομαι ιδιαίτερα. Νομίζω ότι έχει περισσότερο συμφέρον από όλους ε, η δική σας χώρα για την οικονομική ε, ολοκλήρωση, για τη διευκόλυνση αυτή των πληρωμών. Η χώρα σας έχει βάσεις, έχει θεμέλια και πρέπει να τα εμπιστευτούμε τα θεμέλια που έχετε για να βγείτε από την κρίση. Και σίγουρα και εμείς πρέπει να κάνουμε προσπάθειες αλληλεγγύης και τις κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά όταν δει κανεί ε, τα θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία τη Ελλάδα, ιδίω ό,τι αφορά την τουριστική υποδοχή, την τουριστική ανάπτυξη και τι ανταλλαγέ, βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι μία από τι χώρε που πραγματικά έχει ίσω και το μεγαλύτερο συμφέρον να υπάρχει η μεγαλύτερη ολοκλήρωση ε, τη ε, ενία αγορά. Ένα άλλο θέμα το οποίο εθίγει είναι για τι κανονικέ πληρωμέ και αναλήψει. Έχουμε προβλέψει ε, κάποια πράγματα. Κύριε Μάρτιν, τώρα κατά πόσον μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Κοιτάξτε, εγώ έχω δεσμευτεί προσωπικά να μελετήσω το θέμα αυτό ε, και στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για τις πληρωμές και τις επιπτώσεις. Κύριε Κοζές, ο συνήθως έβαλε ο κύριος Κοζές ε, τα σωστά ερωτήματα. Έχουμε και την Πολυμερή Επιτροπή. Θα βρούμε λύση, πιστεύω, ισορροπημένη με τις προτάσεις που θα υποβάλουμε. Συγγνώμη, για τις προμήθειες, για τις δεκρατικές προμήθειες. Αυτές θα προσπαθούμε να τις μειώσουμε. Βέβαια, αναγνωρίζει το κείμενο κύριε Γκοζές ότι η απαγόρευση των πολυμερών αυτών προμηθειών, των καταποκοπή προμηθειών που εφαρμόζουν έξι χώρες, μπορεί να αποτελεί ένα πρόβλημα. Εξού και έχουμε προβλέψει αυτή τη μεταβατική περίοδο. Μέχρι το 2017. Δεν μπορώ να προδικάσω τι θα γίνει βέβαια σε καμία περίπτωση. Σε ό,τι αφορά και τις, τις ε, τραπεζικές κάρτες. Δεν μπορώ να προδικάσω. Το κύριο Μόλιτσερ, ο οποίος ανέφερε τον κανονισμό για τους καταναλωτές και την ασφάλεια, την προστασία που οφείλουμε να εξασφαλίσουμε για τους καταναλωτές. θέλω να σας πω ότι θα ενισχυθούν με τον κανονισμό τα δικαιώματα των καταναλωτών, ώστε να μπορούν ε, να εφαρμόζονται κάποια αυτόματα πλαφών και θα υπάρχουν και ε, ρήτρε προστασία και διατάξει προστασία. Θα πρέπει λοιπόν σε κάθε ε, χρέωση να επιβεβαιώνεται και να επαληθεύεται τι γίνεται για να μην υπάρχει κάποιο δικαίωμα ίσως επιστροφής. Ίσως ήταν λίγο πολύπλοκα αυτά που είπα, αλλά αυτό που θέλω να πω ουσιαστικά είναι ότι προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την προστασία των καταναλωτών. Αν κατάλαβα καλά αυτό που ρώτησε ο κύριος Στογιάνοφ για τις εσωτερικές χρεώσεις, δεν έχω ε, αυτή τη στιγμή ε, στοιχεία για να σας απαντήσω, οπότε θα σας δώσω εγγράφος την απάντησή μου. Πάσκα, Μπασέσκου, Σιλβέστρης και οι τρεις ε, είπαν ε, ότι θα υπάρξουν μεγάλες εξοικονομήσεις και για τους ε, καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις και έχουν δίκιο. Επίσης, κυρία Μπένοβα μίλησε πόσο ευνοϊκό θα είναι αυτό το πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα. Δίκιο έχει και η κυρία Μπένοβα. Να ευχαριστήσω τέλος τον κύριο Κάρα ο οποίος τόνισε την προστιθέμενη αξία, που είναι και το τρίτο σημείο που συζητούσαμε και πριν για την προσθέμενη αξία της εσωτερικής αγοράς. Θέλω να πω όπως και ο κύριος Κάρας, να πω και στον κύριο Ζέμκε, ότι το σχέδιο αυτό αφορά όλες τις πληρωμές ευρώ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο τις χώρες της Ευρωζώνης. Επαναλαμβάνω, ε, αφορά όλες τις χώρες που ε, πραγματοποιούν πληρωμές ευρώ εντός της Ένωσης και όχι μόνο αυτές που είναι αυτή τη στιγμή ε, στο ευρώ. Θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά ολοκληρώνοντα ε, την εισηγήτρια για την πολύ ποιοτική τη έκθεση. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση γύρω από την έκθεση Σάρι Εσάγια ολοκληρώθηκε. Σα ενημερώνω ότι η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στι 12 το μεσημέρι. Το επόμενο θέμα στην ε, ημερήσια διάταξη είναι προφορική ερώτηση προ την Επιτροπή για τη συλλογική διαχείριση